και θα πάρουμε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, η συζήτηση να γίνει στις 5 και μισή περίπου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις να θεωρηθεί δεκτή η πρόταση αυτή. Πρόεδρε, δεν θα ήθελα να ζητήσω να έρθει κάποιος από την Ισραηλινή αντιπροσωπεία, μόνο πρέσβης. Είναι απαράδεκτο για μας το Ισραήλ και η αντιπροσωπεία του Ισραήλ να μας στέλνει ε, κατωτάτου επίπεδου διπλωμάτες για τη συζήτηση αυτή. Πριν φτάσουμε στο συγκεκριμένο θέμα συζήτησης, θα ήθελα να συμφωνήσουμε όλοι για το να γίνει η συζήτηση στις 5.30 ή γύρω εκεί στις 5.30 το απόγευμα. Λοιπόν, συμφωνείτε όλοι. Δεύτερον, η κυρία Άστον, όπως είπα, δεν είναι διαθέσιμη. Συμφωνείτε να ζητήσουμε από τον πρόεδρο του ΚΟΠΣ να είναι παρόν στις 5 και μισή. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις γύρω από αυτή την πρόταση. Το τρίτο σημείο πάνω στο οποίο θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση είναι η παρουσία κάποιου, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος, από την Ισραηλινή αντιπροσωπεία. Ο συνάδελφος που μόλις πήρε το λόγο είπε ότι ε, δεν συμφωνεί για την παρουσία του πρέσβη. Όχι λέει ο κύριος Βάιγκελ, παρανόηση. Εγώ ακριβώς αυτό είπα είναι να είναι παρόν ο πρέσβης, όχι κάποιος κατωτέρω επίπεδο. Μόνο ο πρέσβης. Λοιπόν, θα πρέπει να πάρουμε απόφαση για την παρουσία του πρέσβη του Ισραηλινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, σωστό είναι αυτό που λέει ο συνάδελφος. Όχι όποιος να είναι από την Ισραηλινή πρεσβεία. Πρέπει η Επιτροπή μας να δώσει βάση στο να έρθει ο... κάποιος τουλάχιστον από την Ισραηλινή πρεσβεία, οπότε θα μπορούσε να είναι κάποιος ε, πλήρεξούσιος ε, υπουργός ή κάποιος τέτοιο βαθμού. Κύριο Σαλαφράγκα, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το επίπεδο επικοινωνίας ε, το οποίο θα πρέπει να έχουμε γύρω από το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιστοιχεί ε, στην παρουσία του πρέσβη ε, ε, της πρεσβείας του Ισραήλ και όχι της αντιπροσωπείας του Ισραήλ και όχι ενός απλού εκπροσώπου, ενός απλού υπαλλήλου. Γιατί αν είναι να έρθει ένας απλός υπάλληλος να μην γίνει μια τέτοια συνάντηση. Και καταρχάς συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Σβόμποντα, ας αναβάλουμε την ψηφοφορία για την Αλβανία και ας περιμένουμε να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. για τη συνάντηση με το Ισραήλ. Έχει σημασία να συναντηθούμε με τον ίδιο τον πρέσβη του Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά από αυτά τα οποία προηγήθηκαν της αναχώρησης της αντιπροσωπείας μας στο Ισραήλ και των πιέσεων που υπέστημεν από τον πρέσβη του Ισραήλ. Πρέπει να είναι ο ίδιος παρόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν και εγώ μέλος αποστολή στο Ισραήλ. Είχαμε μια συνομιλία και με τον κύριο Άγελον. Ξεκαθαρίσαμε πως η συμπεριφορά του πρέσβη πριν από το ταξίδι μας δεν ήταν αυτή η οποία περιμέναμε και εγώ θεωρώ πως πρέπει να έρθει εδώ πέρα ο πρέσβης πρέπει να μιλάμε με τον υψηλότερο εκπρόσωπο του Ισραήλ να μπορεί να μας πει ότι είναι και βεβαίως ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα καθώς δεν είναι εδώ πέρα και ο κύριος Αλμπερτίνη σήμερα. Κάτι άλλο ακόμα λένε πως ε, θα γίνει εδώ πέρα μια υποδοχή του κυρίου Μωτάκη σε μια δεξίωση στην οποία θα σερβιριστεί κρασί. Μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Δεν το βρίσκω σωστό αυτό. Ε, ε, Καλώ συνάδελφοι, εγώ θεωρούσα δεδομένο ότι η αντιπροσωπεία του Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη. Πέραν αυτών και μετά από όσα προηγήθηκαν, προβλέπετε λοιπόν από εδώ και πέρα στις 5.30 μετά τις ψηφοφορίες η συζήτηση γύρω από τη Γάζα. Θα έχουμε τον πρόεδρο του Κόψ και θα ζητήσουμε επίσης ε, και την παρουσία μόνο του Ισραηλινού πρέσβη. αν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, για την υιοθέτηση των πρακτικών της 14ης Απριλίου και της 4ης Μαΐου. Έχετε το λόγο κύριε Χουντή. Δεν πήρα το λόγο για τα πρακτικά σας ζητώ επανειλημμένα το λόγο για μια διαδικαστική πρόταση που κατατέθηκε και δεν ξέρω επειδή είμαι πίσω δεν με βλέπετε δεν μου δώσατε το λόγο. Ετέθη στην ημερήσια, πρόταση στην ημερήσια διάταξη αν θα γίνει η ψηφοφορία για την Αλβανία. Και σας ζήτησα το λόγο επειδή είμαι ο εισηγητής. Δεν έχω αντίρρηση να την αναβάλουμε αυτή την συζήτηση εφόσον περιμένουμε ε, και την ψηφοφορία εφόσον περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Αν αυτό πιστοποιηθεί, δεν κατάλαβα αν πράγματι εγκρίθηκε αυτή η πρόταση με συμφωνία όλων, τότε θα προσδιορίσει και τη δική μου εισηγητική παρουσίαση στη συζήτηση που θα γίνει. Γιατί θα... Ναι, λέω, συμφωνώ να γίνει η αναβολή, την πρόταση που έκανε ο κύριος Σβόμποντα όσον αφορά την ψηφοφορία, ελπίζοντας ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις ε, αισιόδοξε, κατόπιν τούτου να ξέρω κι εγώ πού θα κινηθεί η παρουσίαση που θα γίνει στη μετέπειτα διαδικασία. Αυτό σας παρακαλώ διευκρινίστε. Inizieremo adesso Inizieremo adesso il dibattito sull'Albania e quindi lei avrà ovviamente tutte le possibilità. Λοιπόν, ε, προσπαθούμε να δούμε όλες τις δυνατότητες ε, τι οποίε έχουμε πριν πάρουμε απόφαση. Λοιπόν, όταν έρθει η στιγμή θα αποφασίσουμε ακριβώ τι θα πρέπει να γίνει. Diamo per approvato quindi il processo verbale del... Θεωρούνται δεδομένα τα πρακτικά της 14ης Απριλίου και της 4ης Μαΐου και ξεκινάμε αμέσως τη συζήτηση της πρότασης ψηφίσματος για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας. Είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Έχουν κατατεθεί 114 τροπολογίες στο κείμενο του εισηγητή, του κ. Χουντή. και μιας και κανονικά προβλέπεται η ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα και για να διευκολύνει την ψηφοφορία ο εισηγητής σε συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές προετοίμασε εννέα συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να δώσω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή αμέσως για να μας μεταφέρει τις απόψεις του και να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ε, δεν θα ναι, ναι, επαναλάβω τις βασικές διαπιστώσεις και προτάσεις που κάνει το ψήφισμα. Στο μεσοδιάστημα έγινε προσπάθεια με τους σκιώδεις ε, εισηγητές των άλλων πολιτικών ε, ομάδων να βρεθούν συμβιβαστικές λύσεις. Νομίζω ότι έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους διότι συνέβαλαν στο να διαμορφώσουμε συμβιβαστικές προτάσεις ε, συντομεύοντας αν θέλετε και περιορίζοντας τις επιμέρους τροπολογίες πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια και ότι καταφέραμε σε αρκετά σημεία να έχουμε συμβιβαστικές προτάσεις εκφράζει κατά βάση έτσι θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι θα φανεί και στην τελική ψηφοφορία ότι στις βασικές εκτιμήσεις, στις βασικές προτάσεις είμαστε ε, λέω κατά βάση σύμφωνοι και επομένως λίγα είναι τα ζητήματα που θα μπορούσαν να είχαν, ας το πούμε έτσι, διαφορετικές απόψεις ή που να έδιναν περαιτέρω, ας το πούμε, συζητήσεις. Επομένως, εγώ θα σταθώ σε δύο-τρία θέματα που έχουμε σε σχέση με τις εξελίξεις και με το ζήτημα που κουβεντιάσαμε. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρώτο θέμα, κεντρικό ζήτημα, στην έκθεση και αν θέλετε και στην πορεία, την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας είναι η λύση της πολιτικής κρίσης, η άρση του σημερινού πολιτικού αδιεξόδου. Είναι κεντρικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να το παρακάψει κανεί. Εκεί έγιναν και περισσότερε τροπολογίε. Εκεί έχει υπάρξει μια νομίζω σωστή συμβιβαστική πρόταση. Έχουμε τι εξελίξει αυτών των ημερών. Υπάρχει, επέστρεψε η ομάδα της αντιπολίτευσης στα έδρανα του Κοινοβουλίου, αλλά παραμένει ω εκκρεμότητα η ερμηνεία και η αποδοχή των εκλογικών αποτελεσμάτων των εκλογών του Ιουνίου έκλεισε ένας χρόνος. Πιστεύω ότι ας ελπίσουμε πια ότι αυτές οι συνομιλίες ενδεχομένως δώσουν κάποια λύση, μακάρι να δώσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα. Προς το παρόν όμως, παρά την είσοδο της αντιπολίτευσης στη Βουλή, το αδιέξοδο όσο αφορά αυτή την ερμηνεία παραμένει και επομένως η ένταση δεν έχει πέσει. Άρα και η πολιτική κατάσταση έχει μια σχετική, ε, είναι εύστραστη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που θα ήθελα να πω. Το δεύτερο έχει να κάνει με την υπόθεση της απελευθέρωσης της βίζας, της απελευθέρωσης της βίζας. Εξ όσων γνωρίζω, η Επιτροπή έκανε δεκτή την πρόταση στις 27 Μαΐου και προχωράει εξετάζοντας εκκρεμή στοιχεία να διατυπώσει μια νεότερη υποθέτω θετική πρόταση για την Αλβανία και για τη Βοσνία και η Ερσεγοβίνη και επομένως αν έτσι είναι τα πράγματα και νομίζω πως είναι έτσι, να το χαιρετήσουμε και νομίζω ότι στην έκθεσή μας, στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, πρέπει να μείνουμε παρά τις όποιες παρατηρήσεις που θα μπορούσε να κάνει κανείς, αλλά συνδέοντάς το με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση, να παραμείνουμε επί της θέσης αυτής αρχής ότι οι Αλβανοί πολίτες έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και αυτοί ελεύθερα και επομένως να προτρέπουμε για να αντιμετωπιστεί αυτό το, το θέμα. Στα άλλα ζητήματα, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να πω πολλά. Υπάρχουν οι τροπολογίες, υπάρχουν οι συμβιβαστικές προτάσεις. Ελπίζω και με τη συζήτηση να τα προσεγγίσουμε καλύτερα τα θέματα. Ε, νομίζω ότι εν τέλει από την έκθεσή μας θα πρέπει να παραμένει ζωντανή η προπτική και το κίνητρο όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κίνητρο για να προχωρήσουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και για να προχωρήσουν σε βελτιώσεις σε όφελος των πολιτών τους και βεβαίως σε όφελος της ειρήνης και της ασφάλειας. Αυτή είναι η μέρημνα και η κεντρική κατεύθυνση της έκθεσης. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι συμβιβαστικές προτάσεις. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ τους κοιόδους εισηγητές για τη συμβολή σε αυτή την ε, προσπάθεια και τη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί συνεχίζει να μας βοηθάει ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Grazie. Allora, i relatori ombra sono... Σκιώδης εισηγητές. Πακ, Σβόμποντα, Σαρτζεντίνη, Σάκε. Με τη σειρά μπορούν να πάρουν το λόγο πρώτη η κυρία Πακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τον κύριο Χουντή είχαμε μία ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη συζήτηση με τις, για τις πολλές τροπολογίες και συμφωνήσαμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Εντάξει, μπορεί να είναι μια κάποια με την οποία δεν συμφωνώ, αλλά όλες τις νέες μπορούμε να τις εγκρίνουμε από κοινού. Επίσης ε, για το θέμα της εκπαίδευσης ε, δόξα το Θεό ε, αποδόθηκε περισσότερη σημασία με δύο τροπολογίες από ό,τι μέχρι στιγμής και είναι σημαντικό αυτό για όλη την περιοχή, ειδικά το ότι αυτές οι χώρες μπορούν να συμμετέχουν στα δικά μας προγράμματα ε, τα εκπαιδευτικά. Αυτό σημαίνει όμως πως πρέπει να έχουν υπηρεσίες που να μπορούν να τα διαχειριστούν αυτά τα πράγματα. Οπότε μια τέτοια όθηση είναι σωστή. Εντάξει, συμφωνώ με την αναβολή, αλλά η έκθεση αυτή, όπως έχει, δεν θα αλλάξει και μετά από μια συμφωνία στην Αλβανία. Το πολύ πολύ να α, λείπει μια παράγραφος, γιατί θα έχει λανθασμένα γεγονότα τότε. Αλλά εάν δούμε την Αλβανία πρέπει να δούμε λίγο τα γεγονότα δεν πρέπει να συμπεριφερθούμε διαφορετικά από ότι έναντι μια άλλη χώρα. Εγώ παρακολουθώ την ε, κατάσταση στην Αλβανία εδώ και 20 χρόνια και πάντα προσπαθούσα να μην μεροληπτώ και όταν ήταν ο Μπερίσα στην αντιπολίτευση και στην ε, κυβέρνηση και δεν συμπεριφέρονταν όπως περιμέναμε από ένα δημοκρατικό κράτος ασκούσα κριτική πάντα δημοσίες. Οπότε κανείς δεν μπορεί να μου πει πως κάποτε μερολήπτησα. Πρέπει να πω μόνο πως αυτά τα οποία ζούμε τώρα είναι πράγματα τα οποία δεν, δεν επιτρέπονται σε μια δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει ένας εκλογικός νόμος ο οποίος πριν από δύο χρόνια και η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση έκαναν εκλογικό νόμο στον οποίο βασίζονται αυτές οι εκλογές. Και ήταν οι πρώτες εκλογές οι οποίες ήταν αυτές οι οποίες μέχρι τώρα πήγαιναν προς κάποια ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για πρώτη φορά. Μετά τις εκλογές και οι σοσιαλιστές παρατηρητές των εκλογών δεν έφεραν κάποια αντίρρηση στις εκλογές. Οι, παρατη... οι αντιρρήσεις έγιναν όταν σχηματίστηκε κυβερνησία κυβέρνηση ένα, από ένα άλλο σοσιαλιστικό κόμμα με αυτό το δημοκρατικό κόμμα. Εγώ το ε, έβρισκα θετικό το ότι είναι δυνατόν σε μια χώρα όπως η Αλβανία που δεν έχει τόσο μεγάλη δημοκρατική παράδοση δύο πόλοι να συμφωνήσουν να κατευθυνθούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ το χαιρέτησα. Αυτό βεβαίως δεν το χαιρέτησε η αντιπολίτευση, μποϊκοτάρισε και το κοινοβούλιο. Τον Μάρτιο προσήλθαν στο κοινοβούλιο γιατί θα έχαναν τις εντολές τους, αλλά τις έδρες τους, αλλά δεν εργάστηκαν τακτικά και μετά ξεκίνησε μια απεργία πείνας. Ε, τι γίνεται δηλαδή εδώ πέρα. Αν η αντιπολίτευση διαπιστώνει λάθη στην εκλογική διαδικασία μπορεί να πάει είτε στο συνταγματικό δικαστήριο είτε να προσβάλλει τη διαδικασία αλλά δεν μπορεί να απαιτεί αυτά τα οποία απαιτεί από την κυβέρνηση πρέπει να τηρούμε αυτό δεν το κάνουμε πουθενά ούτε εμείς τηρούμε την νομοθεσία, την εκλογική νομοθεσία. Αν θέλουν να φέρουν κάτι στο δικαστήριο, να το κάνουν. Ε, κατά την άποψή μου αυτό είναι το μόνο σωστό το οποίο μπορεί να γίνει. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μην υποστηρίξει καμία ομάδα εδώ μέσα κάτι το οποίο δεν στέκει σε καμία άλλη χώρα. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από μια χώρα και μία κυβέρνηση να παραβιάσει τους νόμους και το σύνταγμά της. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να βοηθήσουμε τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, να τους προσφέρουμε κάποιες δυνατότητες να συζητήσουν για αλλαγές στον εκλογικό νόμο ή στον ε, κανονισμό του Κοινοβουλίου για το μέλλον ή για τις επόμενες εκλογές που έρχονται ή τις δημοτικές αλλά να μην πάρουμε το πλευρό τη μίας πλευράς, να δούμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι όπως σας τα περιέγραψα, δεν είναι μόνο μερι. Έτσι είναι. Γι' αυτό παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να πείσουν τα κόμματα εκεί επιτόπου, να κοιτάξουν προς το μέλλον, να δημιουργήσουν κανόνες για το μέλλον, αλλά όχι για το παρελθόν. και θα πρέπει να έρθει και η αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο γιατί ορισμένα πράγματα μπορούν να κανονιστούν μόνο με μεγάλες πλειοψηφίες στο, στο κοινοβούλιο. Και είναι πράγματα επίσης τα οποία είναι σημαντικά και για την πρόοδο τους προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Βόμποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά του και συμφωνώ με την κυρία Πακ πως ε, στα περισσότερα πράγματα δεν θα αλλάξει πράγματι τίποτα, είτε στην κριτική, είτε στις προτάσεις, είτε σε αυτά τα οποία προτείνουμε. Στην Αλβανία έχει κάνει πρόόδο η Αλβανία, πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και θέλουμε περισσότερη πρόοδο, να υπάρχει και εσωτερική ειρήνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε απελευθέρωση της ε, βίζας για να ξεκινήσει μια δικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακριβώς επειδή λοιπόν ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για την πρόοδο της ε, Αλβανίας, είναι κατά την άποψή μου σωστό να προσπαθήσουμε και να βρούμε μία συνένεση. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα να αναβάλουμε, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να ψηφίσουμε πριν τις διακοπές του καλοκαιριού, γιατί είχαμε προγραμματίσει και πρέπει να ξέρουμε πως το αργότερο για να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια είναι ο Ιούλιος. Και αυτό πρέπει να γίνει. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε προς το τέλος η κυρία Πακ, αλλά δεν θα ήθελα τώρα εγώ, όπως έκανε η κυρία Πακ, να κατανείμω τις ευθύνες. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είχε αναγνωριστεί ως νόμιμη και από την αντιπολίτευση, αυτό δεν αλλάζει. Αλλά υπάρχουν παρατηρήσεις όσον αφορά πιθανές βελτιώσεις στον εκλογικό νόμο και το θέμα είναι ποια είναι τα βήματα για να επιτευχθεί αυτό. Τα δύο κόμματα έχουν ξεκινήσει ε, συνομιλίες γιατί εμείς ως σοσιαλδημοκράτες και το ΕΛΚ μιλάνε και είπαμε εμείς στα αδελφά μας κόμματα πως πρέπει να καταλήξουν σε μια λύση οπότε έχουμε τη συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού του κ. Μπερίσα και της αντιπολίτευσης. Κάποια πράγματα έχουν ε, γίνει. Υπάρχει συμφωνία για την σύσταση μιας ειδική επιτροπής στο Κοινοβούλιο όπου θα ορίσει τον πρόεδρο η αντιπολίτευση και θα έχει την πλειοψηφία, αλλά η διαδικασία και εντολή αυτής της επιτροπής δεν έχει ακόμα καθοριστεί, οπότε το θέμα, όπως είπαμε, δεν είναι αλλαγή του αποτελέσματος των εκλογών, απλά να αλλάξει η νομοθεσία για τις μελλοντικέ εκλογές. πολύ ε, και η κυρία Πάκα ε, και εγώ που ασχολούνται χρόνια με αυτό το θέμα, βλέπουμε πως είναι δύσκολο να επιτευχθεί συνένεση αν και πράγμα το αναγνωρίζουμε πως οι τελευταίες εκλογές ήταν καλύτερες από άλλες στο παρελθόν. Αλλά βεβαίω πρέπει να γίνει ακόμα αρκετή πρόοδος. Ευχαριστούμε επίσης τον εισηγητή για την διάθεσή του να δεχτεί μια αναβολή. Όπως σας είπα όμως το αργότερο όριο πλέον είναι ο Ιούλιος Νομίζω πως ευθύνη μας ε, είναι πράγματι να βρούμε κάποιες ε, συνενέσεις. Πρέπει λοιπόν να γίνουν αυτά τα τελευταία βήματα γιατί όπως είπαμε το επόμενο μήνυμα θα ήταν η απελευθέρωση της βίζας την οποία θα θέλαμε να, να δώσουμε αλλά πρέπει να υπάρξει και μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σβόμποντα. Ο κύριος Σαρτζεντίνη και μετά ο κύριος Κασίν. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω όπως ε, και ο Στίβεν Χιούς. επανήλθε η αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο και η Κομισιόν μιλάει για απελευθέρωση της βίζας. Αυτά είναι θετικά νέα. Τώρα, το να πάει αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αλβανία για να βοηθήσει πράγματι είναι θετικό βήμα, αλλά ας περιμένουμε λίγο και ας περιμένουμε λίγο εδώ πέρα, ενώ να μην ψηφίσουμε σήμερα το πρωί. Επίσης όμως θα πρέπει να γίνει ένα κρίσιμο βήμα πριν τις διακοπές του καλοκαιριού, να στείλουμε δηλαδή το ε, μήνυμα στους ε, Αλβανούς πολίτες, πως εντάξει δυστυχώς θα μπορέσουν να έρθουν διακοπές ως το καλοκαίρι, αλλά από το φθινόπωρο θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα. Επίσης τώρα έχουμε μια νέα πρόταση από τον εισηγητή. Στο σημείο 18 έχουμε τη συμβαστική λύση 5, η αρχική παραγραφός 18. Δεν μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα αναφέρεται ε, επισύρει την προσοχή στην σημασία της απογραφής για όλες τις εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες της απογραφής που προγραμματίζεται για το 2011 για εμάς ε, αυτό είναι αντίφαση με αυτό το οποίο ακολουθεί που μιλάει για την ελεύθερη για τον ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό, δηλαδή να είναι επιλογή του καθενός να πει σε ποια εθνοτική ομάδα νίκη. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον εισηγητή να το ξανασκεφτεί αυτό το σημείο. Επίσης νομίζω πως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ευρύτερες ε, πλειοψηφίες αν δεν ψηφίσουμε σήμερα. Τέλος. Είμαι ικανοποιημένη με το πώς ε, είδε τους ε, συμβιβασμούς ο εισηγητής. Πράγματι είναι πάρα πολύ θετικά όλα αυτά και η ε, διάθεση την οποία επέδειξε. Για τους φιλελευθέρους ο κ. Κασίν. Και εγώ θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες λέγοντας ότι σήμερα δεν πρέπει να ψηφίσουμε. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να περάσουμε και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μετά την επιστροφή της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όλοι περιμένουμε ότι θα συμβεί, γιατί πρώτα-πρώτα θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για τον κύριο Χουντή, γιατί δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και γιατί πάρα πολύ καλά διατύπωσε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος όσον αφορά την ένταξη της Αλβανίας. Επίσης θα πρέπει να χαιρετήσουμε το ότι αυτός ο διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ε, γνωρίζει μια νέα θετική φάση. Είχαμε 19 ε, και 20 Μαΐου αυτές τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, την απεργία πείνας, γιατί ο ρόλος ε, της Κομισιόν και του, και του αρμόδιου επίτροπου έπαιξαν ένα πάρα πολύ θετικό ρόλο τόσο ώστε να μπορέσουμε να απεμπλέξουν την κατάσταση που είχε κρατήσει ένα χρόνο στην Αλβανία αυτή, αυτή την εμπλοκή. Όμως θα πρέπει να καταλήξουν κάποια συμφωνία και όλα όσα έχουν γίνει δείχνουν ότι θα πρέπει να βοηθιέται ο διάλογος και να δίνεται μια όθηση στο δημοκρατικό προτσές ούτως ώστε να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη όλη η περιοχή, γιατί χωρί διάλογο και χωρί πλήρη δέσμευση όλων των πολιτικών πτερήγων του, του Κοινοβουλίου και τη χώρα γενικότερα, η Αλβανία δεν είναι δυνατόν να σημειώσει κάποια πρόοδο και να έρθει στην αγκά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει αυτέ τι προσπάθειε να συνεχιστούν. Θα πρέπει να αποδείξει η Αλβανία στους εταίρους της και στην Ευρώπη ότι μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα σοβαρά της πολιτικά προβλήματα. Όλα τα κόμματα στην χώρα θα πρέπει να βάλουν στην πάντα τις διαφορές τους και θα πρέπει να πρετανεύσει δημοκρατικό πνεύμα και έτσι να, αναζητηθεί μια λύση εις ε, την σημερινή κατάσταση και έτσι θα συνεχίσει η διαδικασία αυτή. Άρα θέλουμε γρήγορα εξελίξεις και θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να μας ε, καθησυχάσει η Αλβανία ότι μπορεί να συνεχίσει αυτή την πορεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κασίν. Άλλοι πέντε συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί έχουμε αργήσει. Σεβερίνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω και μα απασχολεί η υπόθεση σύνταξη τη Αλβανία στην Ένωση. Αυτό είναι το θέμα τη έκθεση. Και βέβαια είναι αυτό σημαντική υπόθεση και για τους αγνούς, αλλά και για μας. Πάντως, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτή μας τη δέσμευση και στους όρους και προποθέσεις που θα ισχύσουν. Οπότε, η, η αναβολή της ψηφοφορίας δεν είναι θέμα διαδικαστικό. Τώρα μας ακούν και μας βλέπουν συνάδελφοι Ελβανοί και πρέπει να τους διαβιώσουμε ότι πρόκειται για μήνυμα και απόφαση πολιτική που στέλνουμε στο, στο, στα τύρανα, ούτω ώστε οι πολιτικέ δυνάμει τη χώρα θα πρέπει να μπορέσουν να συνεχίσουν έναν διάλογο δημοκρατικό, θετικό, ορθολογικό. Και αν δεν μπορούν να το κάνουν, τότε διακυβεύεται η πορεία του προ την Ευρώπη. Όχι, φυσικά και εμεί πρέπει να είμαστε ουδέτερε στι εκεί διαφορέ και προστριβέ και συγκρούσει. Ούτε είναι δυνατόν εμεί να υποκαταστήσουμε τους ε, αρμόδιου δικαστέ. Όμω δεν μπορούμε παρά να διατυπώσουμε το ότι σε κάθε εκλογή στην Αλβανία ακολουθεί μια κρίση εδώ και χρόνια, αν όχι εδώ και δεκαετία. Επομένω, πάει κάτι πάει στραβά με το σύστημα στη χώρα. Και δεν έχει σημασία ποιο ήρξε το χειρόν αδίκο και ποιο φταίει και ποιο δεν φταίει. Στη σημερινή συγκυρία αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα και ότι τα πολιτικά κόμματα στη χώρα δεν είναι ει θέση να εκτονώσουν την κατάσταση. Και ακριβώς αυτό μας προβληματίζει. Οπότε όλοι στη χώρα θα πρέπει να καταλάβουν ότι άπαξ και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την εσωτερική τους κρίση, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν την πορεία τους προς την Ένωση. Εν κατακλείδη, να μην διστάζουμε, συνάδελφοι, να επενέσουμε αυτούς για τόσο κατάφερε η ευρωπαϊκή διπλωματία. το ότι οι σοσιαλιστές συνεπήκαν στο κοινοβούλιο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διπλωματίας μας που στηρίχθηκε και απλώς τις στο κοινοβουλίο και το ότι σταμάτησαν οι απεργίες πείνας ακριβώς και αυτό είναι αποτέλεσμα των διαβημάτων της ε, διπλωματίας μας και το ότι υπάρχει κάποιος διάλογος που συνεχίζεται και αυτό επίσης οφείλεται στις προσπαθίες μας. Άρα εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με το θέμα μέχρι ότου αν βρεθεί μια λύση. Και αν δεν βρεθεί λύση, τότε θα τους πούμε ξεκάθαρα ότι όλα, όλα, όλα τίθενται να αμφιβόλω και πρώτα-πρώτα και οι διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Σύνδεσης και για την ε, κατάργηση της θεώρησης διαβατήριων. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο προ τα τύρανα. Και επίση να του καθαρίσουμε ότι τον μπαλάκι στο δικό του γήπεδο. Από αυτού εξαρτάται τι θα γίνει η χώρα του για τι σχέσει με την Ένωση. Ο συνάδελφο Τάλερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα της Αλβανίας είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ε, άμεσα και έχει διανύσει βέβαια και αρκετά μεγάλη απόσταση η Αλβανία μετά από τις τρομερές πολιτικές αλλαγές εδώ και αρκετά χρόνια. Βέβαια το βασικό χαρακτηριστικό της αλβανικής πολιτικής σκηνής είναι η μη επικοινωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση κάθε φορά. Έτσι ακριβώς αυτή η μη επικοινωνία δεν μπορεί να μας οδηγήσει κάτω από τις παρούσες συνθήκες σε μια λύση του πολιτικού προβλήματος. Καταδικάζει τους δύο πολιτικούς σχηματισμούς σε μόνιμη αντιπαράθεση. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, όπως είπε ο κύριος Σεβερίν, και σε επίπεδο πίεσης από πλευράς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Επιτρόπου Φούλε για να ξεπεραστούν αυτές ε, οι αντιθέσεις. Θα πρέπει και η αλβανική δημοκρατία να αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ξεπεραστούν κάποιες προσωπικού τύπου αντιπαραθέσεις μια επιθετική ρητορική η οποία λειτουργεί αρνητικά για την πολιτική συνοχή της χώρας και παραλαμβάνω ότι αυτό αφορά και τους δύο μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς, όχι μόνο ε, την κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τα τύρανα, να δείξουμε ποιες είναι οι προσδοκίες τις οποίες έχουμε. Περιμένουμε η δημοκρατία να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να επιτρέψει στην Αλβανία να λειτουργήσει σωστά, χωρίς βίζες, κάτι το οποίο ενδιαφέρει τόσο πολύ τον αλβανικό λαό. Κυρία Σήμερα η κατάσταση στην Αλβανία είναι ακόμα πολύ κρίσιμη και αυτό ε, το μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα που παρατηρούμε σήμερα μας δείχνει ότι στην περίπτωση της Αλβανίας είχαμε βιαστεί να θριαμβολογήσουμε τα προηγούμενα χρόνια για την πρόοδο στον τομέα αυτό, ενώ υπήρχαν σοβαρά προβλήματα σε όλες τις εκλογές, όπως αναφέρθηκε από πολλές συναδέλφους, τα οποία τα γνωρίζαμε. Ε, η κίνηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο σημαντικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, έπαιξε πάρα πολύ θετικό ρόλο γιατί πραγματικά νομίζω πριν 15 μέρες η κατάσταση ήταν ε, στα όρια να τεθεί εκτός ελέγχου και να μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα και για περίπτωση έκρηξης βίας. Η έκθεση του κύριου Χουντή είναι μια σωστή και έντιμη αποτύπωση της κατάστασης στην Αλβανία ε, και των ε, μέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν στο μέτρο. Η αναβολή της ψηφοφορίας θα δώσει νομίζω το σωστό μήνυμα το οποίο πρέπει και θα επιτρέψει να ε, ολοκληρωθεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στην περιοχή. Έχει σημασία νομίζω να τονίσουμε και όπως διαφαίνεται από τη συζήτηση είναι καθαρό ότι υπάρχει κοινή ευθύνη των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων στην Αλβανία για τη σημερινή κρίση. Κανείς δεν είναι αθώος του αίματος θα έλεγα για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση και όλοι πρέπει να δείξουν, ε, να καταβάλουν προσπάθειες ώστε η χώρα να ξαναμπεί στον δημοκρατικό δρόμο. Όσο αφορά το θέμα της βίζας νομίζω είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Ε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τιμωρηθούν οι πολίτες για τα μεγάλα ελλείμματα των ηγεσιών τους, των ηγεσιών των πολιτικών κομμάτων αλλά παρόλα αυτά το θέμα της αιρεσιμότητας όπως το έθεσε και ο κύριος Σεβερίν νομίζω έχει μεγάλη σημασία να εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ. L'onorevole Madlener, prego. Madlener. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε. Το Κοινοβούλιο βεβαίως θα πρέπει να συνεισφέρει στην καλύτερη ε, στην καλτέρευση των ε, ζώων των χωρών της Ευρώπης. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για την Αλβανία, για τόση οργανωμένη εγκληματικότητα που μιλάμε για ένα κράτος μαφία και μιλάτε εδώ πέρα για απελευθέρωση της βίζας για να έρθουν πιο εύκολα αυτοί οι εγκληματίες στις χώρες μας. Επιπλέον είναι μια Ισλαμική χώρα το Ισλάμ δεν είναι μια απλή θρησκεία, είναι μια ιδεολογία και αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην Ευρώπη. Δεν αντιλαμβάνω γιατί ασχολούμαστε για να έρθουν αυτές οι φτωχές διεφθαρμένες χώρες στην Ευρώπη. Πραγματικά το βρίσκω ακατανόητο το πώς εξυπηρετούμε τους πολίτες μας με τις αποφάσεις που λαμβάνει αυτό εδώ το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ultimo intervento, la collega η κυρία Γιαννάκου τελευταία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ προσεγμένη εκθεσή του η οποία εν περιλαμβάνει ε, όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία της δημοκρατίας στην Αλβανία. Ε, κύριε Πρόεδρε, η Αλβανία είναι βέβαια... Εγώ προσωπικά ασχολούμαι από διάφορες θέσεις τα τελευταία 20 χρόνια με την Αλβανία. Είναι και μια ιδιότυπη κατάσταση που αφορά ε, στις εσωτερικές φυλές θα μπορούσα να πω που υπάρχουν στην Αλβανία και στις αντιλήψεις που διακινούνται στο νότο και στο βορρά. Ωστόσο το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί από τη συγκεκριμένη αντιπολίτευση. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποχωρεί από τη Βουλή. Νομίζω αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς και αυτό εν συνεχεία, δηλαδή το ποιο ευθύνεται ας το αποτιμήσουν οι πολίτες της Αλβανίας, είναι πράγματι να καθυστερήσουμε, δηλαδή να μην ψηφίσουμε σήμερα την έκθεση, να δούμε τι θα πούν οι εκπρόσωποι μας οι οποίοι είναι στην Αλβανία αλλά κυρίως ως Κοινοβούλιο να δώσουμε ένα μήνυμα ε, ότι και το θέμα της βίζας δεν μπορεί παρά να εξαρτάται από τη λειτουργία της δημοκρατίας και από την προσπάθεια που γίνεται να αντιμετωπιστεί ε, το οργανωμένο έγκλημα το οποίο όντως διασπείρεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Βέβαια εμείς στη χώρα μας έχουμε πάρα πολλούς Αλβανούς εργαζομένους που είναι σωστοί, που συνεισφέρουν ε, στην οικονομία της Ελλάδος και δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ε, τα προβλήματα μαφίας και λοιπά ξεκινούν από την Αλβανία. Είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες. Έχει μέλλον η Αλβανία όπως όλα τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρώπη ε, αλλά το μέλλον αυτό πρέπει να εξαρτηθεί από τους ίδιους κύριε Πρόεδρε και το μήνυμα πρέπει να είναι πάρα πολύ σκληρό και πάρα πολύ σαφές ότι και η αντιπολίτευση οφείλει να αντιδρά μέσα στο Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση οφείλει να συνεννοείται και να διαβουλεύεται με όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν δώσουμε για την τελευταία λέξη το λόγο στον εισηγητή, θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της αντιπροσωπείας της διακοινοβουλευτικής μας, τον κύριο Κούτσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Δεν θα με ακρηγορήσω γιατί ήδη καλύφθηκα ε, στα περισσότερα που ήθελα να πω και εγώ πρώτα πρώτα. Ένα μεγάλο μπράβο να πω στον εισηγητή μας τον κύριο Χουντή γιατί έδειξε πάρα πολύ καλή διάθεση και καλή πίστη στη συνεννόηση του με τις άλλες πολιτικές ομάδες, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Βέβαια δεν τα πήγαμε ε, άριστα, δεν τα βρήκαμε σε όλα, αλλά ήταν πολύ καλές οι προσπάθειες και νομίζω ότι η αναβολή της ψηφοφορίας, το ότι δεν θα γίνει δηλαδή σήμερα το απόγευμα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οι Αλβανοί να το κλάβουν όχι σαν διαδικαστικό θέμα, αλλά σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πολιτικό υπέρ τους. Θα πρέπει επομένω να εκμεταλλευτούν αυτήν την απόφαση με τρόπο ορθολογικό. Τώρα, έχουμε κάποιες πρόσφατες πολιτικές κινήσεις προς την εξέβρεση κάποιες λύσεις και απεμπλογής από τη σημερινή κατάσταση ούτω ώστε τελικά να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο είδου εγγυήσει για μακροπρόθεσμη πολιτική σταθερότητα και εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. Αυτό περιμένουμε, αυτό προσδοκούμε. Άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε, να έρθουμε αρρωγή σε όλε τι πολιτικέ δυνάμεις τη Αλβανία, Άκουσα τα όσα αναφέρθηκαν, γιατί νομίζω ότι όλοι ειλικρινά θέλουν η Αλβανία να πάρει το δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει και αυτή στην υπόθεση ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και επ' αυτέ τη βάση θα πρέπει να διερευνηθεί μία εξέβρεση λύση. Εγώ και συμφωνώ με την Τόρι Πακ. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία όσον αφορά το τι έγινε στι εκλογέ και το αποτέλεσμά του και υπάρχουν περιθώρια να έχουμε καλύτερη διοργάνωση εκλογών στο μέλλον. και όπως είπε και ο Αντριάν Σέβερη, να μην ξανά έχουμε τέτοια φαινόμενα. Υπάρχει κάτι άλλο σοβαρό. Αυτές οι προϋποθέσεις που έχουν ταχθεί από πολιτικής πλευράς, ε, το πιο αποτελεσματικό του ώστε να πιέσει κανεί είναι αυτή η μέθοδος και ευτυχώς που σήμερα δεν ψηφίζουμε. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το θέμα του τι προϋποθέσεις θα τάξουμε. Τα είπαμε με την κυρία Μάλστον και με τους άλλους επιτρόπους. Δηλαδή να μην πιέσουμε όσον αφορά την κατάρριξη των θεωρήσεων διαβατήριων. Αλλά να χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια τα οποία είχαν υιοθετηθεί και να κάτσουμε και να κρίνουμε πότε θα δώσουμε το πράσινο φως όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και παράλληλα να προχωρήσουμε και στην απελευθέρωση των διαβατήριων και των θεωρήσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή η πολιτική προσπάθεια να συνεχιστεί και από το Κοινοβούλιο και από την Κομισιόν και ελπίζουμε ότι η Αλβανία θα συνεχίσει η τη, στην οποία θα συμμετάσχουν όλε οι πολιτικέ δυνάμει και να καταλάβουν όλοι ότι είναι το μέλλον τη χώρα το οποίο διακυβεύεται. Θα πρέπει να βρεθεί μια οριστική πολιτική λύση που θα διηγήσει σταθερότητα. Λοιπόν, ο κύριος Χουντής για τα συμπεράσματα και κυρίως να μας πει ε, τι θα γίνει για την αναβολή της ψηφοφορίας. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τον προβληματισμό που κατέθεσαν. Ε, νομίζω ότι πρώτον πρέπει να καταλήξουμε, εφόσον φαίνεται ότι όλοι συμφωνούμε, στην αναβολή της ψηφοφορίας, όμως, για να το ξαναπώ άλλη μια φορά, το μήνυμα που δίνουμε προς την ε, πολιτικές δυνάμεις της Αλβανίας με αυτή την αναβολή της ψηφοφορίας είναι να αξιοποιήσουν, να αξιοποιήσουν το επόμενο διάστημα για να βγουν από το πολιτικό αδέξοδο. Ε, διευκρινίζω για άλλη μια φορά ότι η αναβολή που φαίνεται ότι όλοι συμφωνούμε με τις ψηφοφορίες δεν εκφράζει διαφωνίες που δεν, γεφυρώνονται στο επίπεδο της Επιτροπής μας, αλλά εκφράζει τη βούληση όλων μας να δοθεί η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί γρήγορα το αδιέξοδο για να μπορέσουμε να συζητάμε κάτω από άλλους όρους ομαλής κοινοβουλευτικής δράσης και ομαλής κοινοβουλευτικών εξελίξεων. Το δεύτερο το μήνυμα που πρέπει να δίνει η αναβολή είναι εφόσον συνεχίζουμε και από ό,τι φάνηκε στα βασικά να είμαστε σύμφωνοι θα έλεγα να, και από τη δική μου την πλευρά και θα ζητήσω και τη βοήθεια και των άλλων ισκιωδών εισηγητών όπου είναι δυνατόν να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το κείμενο εκτιμώντας ότι τελικά η υπερψήφιση αυτής της έκθεσης δεν θα είναι μια προσωπική ας το πούμε ικανοποίηση μόνο, αλλά θα είναι ένα ακόμα συμπληρωματικό μήνυμα προς τις αλβανικές πολιτικές δυνάμεις, προς την αλβανική κοινωνία, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευρύτατα έχει αρχές, κριτήρια που πρέπει να ικανοποιήσει στην πορεία των αλλαγών και στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνω μεγάλη σημασία, όχι προσωπική, στο ποιο θα είναι το μήνυμα εν τέλει που θα δώσει το, το, το ψήφισμα. Δεν θέλω να επεκταθώ ε, ε, αναλυτικά, κύριε Πρόεδρε, στην πολιτική κατάσταση στην Αλβανία. Θέλω να σα πω ότι την παρακολουθώ έτσι κι αλλιώ και λόγω γειτονία, αφού είμαι από την Ελλάδα, αλλά και λόγω άλλων ενασχολήσεων επί 20 και 25 χρόνια. Έχω τι προσωπικέ εκτιμήσει. Δεν είναι όμω η ώρα. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στο πολιτικό σύστημα. Η έκφρασή του είναι η σημερινή πολιτική κρίση είναι χρόνιες καταστάσεις, με ευθύνη κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά τώρα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας και να βοηθήσουμε και ήδη να αντιληφθούν ότι πρέπει να λυθούν ορισμένα ζητήματα, όχι μόνο για να βγει τώρα από το αδιέξοδο η Αλβανία, αλλά για να έχουμε ορθότερες βάσεις οικοδόμησης ενός ε, δημοκρατικού πολιτικού συστήματος. Και εδώ πρέπει να κάνουν πάρα πολλή δουλειά. Δεν κλείνει το θέμα σε σχέση με το πώ θα βγει το θέμα τη ερμηνεία, τη αποδοχή των εκλογικών αποτελεσμάτων. Αλλά αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα να το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Τέλο, σε σχέση με την απελευθέρωση τη βίζα. Ειλικρινά θα ήθελα να συμμεριστώ και με τις ανησυχίες που έχουν ε, εκφράσει ή που εξέφρασαν και σήμερα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και άλλοι συνάδελφοι. Όμως έχω τη γνώμη ότι σε καμία περίπτωση, μάλλον δεν πρέπει να φανεί ότι η δική μας τάση γίνεται πιο αυστηρή υπό την αίρεση να έχουμε ορθότερες πολιτικές εξελίξεις που θα μπορούσε να ήταν μια σωστή προσέγγιση αλλά να μείνουμε αφού βοηθήσουμε να έχουμε ομαλές πολιτικές εξελίξεις να μείνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση αρχής ότι και οι Αλβανοί πολίτες αφού πληρούν ορισμένα κριτήρια, είναι έτοιμοι όπως έχει υποθεί, θα πρέπει να μην έχουν τη δέσμευση της απελευθέρωσης της βίζας όσο αφορά τις μετακινήσεις. Εν πάση περιπτώσει κύριε Πρόεδρε, πείτε μου ποιο είναι πια το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε θα γίνει η ψηφοφορία και αν της τελικής εν πάση περιπτώσει ψηφοφορίας χρειαστεί μια περαιτέρω συζήτηση που θα σημαίνει να συζητήσουμε τις τροποποίησεις που οι πολιτικές εξελίξεις ενδεχομένως επιβάλλουν σε κάποια σημεία. Αν διαφορετικά δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, να καταθέσω κάποιες τροπολογίες, αν υπάρχουν τέτοιο, παίρνοντα υπόψη και τη συζήτηση στην εξέλιξή της και τις εξελίξεις έτσι όπως θα έχουμε, αν έχουμε και ελπίζω να έχουμε αισιόδοξε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Bene, Καλώς. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που έχω καταλάβει και ε, με αυτά τα οποία αποφασίζουμε, θα ψηφίσουμε στην επόμενη τακτική μας συνάντηση στις 22 και 23 Ιουνίου, εντάξει. Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα αυτό πλέον. Περνάμε τώρα στην κοινή συζήτηση και τα σημεία 6 και 7, όπως είχαμε πει προηγουμένως. για το χρηματοδοτικό μέσο για την πρόθεση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συζήτηση για την τροπολόγηση του μέσου σταθερότητα. σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος που τροποποιεί το Ευρωπαϊκό Μέσο για την πρόθεση της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την τροποποίηση του κανονισμού που προβλέπει την δημιουργία του μέσου σταθερότητας. Σε μια παλαιότερη συνάντηση δόθηκε εντολή στους κυρίους, στην κυρία Μάλλον Γκάλ και στην κυρία Λόχμπίλερ να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται από το 291 σχετικά με τις αλλαγές μάλιστα που συνέβησαν μετά από τη θέση ισχύ της συνθήκης γύρω από τα δύο συγκεκριμένα θέματα. Η ψηφοφορία έχει αναβληθεί αναμένοντας τις τελικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Μετά από πάρα πολλές συναντήσεις και απόπειρες διαπραγμάτευσης δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο που αρνείται να εφαρμοστεί η διαδικασία την οποία ζητά το Κοινοβούλιο. Στις 23 Απριλίου οι συγγήτριες ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις δυστυχώς δεν καρποφόρησαν και πρότειναν με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ψηφίσουμε το σχέδιο ψηφίσματος το οποίο είχε παραμείνει σε εκκρεμότητα γύρω από τα θέματα αυτά. Η ψηφοφορία λοιπόν προβλέπεται να γίνει σήμερα το απόγευμα και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε ταυτόχρονα στην Ολομέλεια και τις τέσσερις εκθέσεις γύρω από τη διαπραγμάτευση αυτή στην Ολομέλεια του μηνός Ιουνίου εννοώ. Θυμίζω ότι μιλάμε για την έκθεση για το μέσο συνεργασία και ανάπτυξη, τη συνεργασία με τις εκβιομηχανοποιημένες χώρες, το μέσο σταθερότητας και το μέσο για την πρόθεση της δημοκρατίας. Αν μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω συνάδελφοι ότι οι τροπολογίες αυτές που έχουν κατατεθεί από τις δύο συνεισηγήτριες σχετικά με την εφαρμογή των συνοδευτικών πράξεων. Μέσω της ψηφοφορίας θα επιβεβαιώσουμε ότι αυτού του είδους η διαδικασία θα πρέπει να εφαρμοστεί και κυρίως για το μέσο σταθερότητας. Η έκθεση για το μέσο σταθερότητας είχε γίνει δεκτή πριν από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Πέρα από αυτά τα εισαγωγικά θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Κίνγκα που είναι η συγγήτρια για το μέσο για την πρόθεση της δημοκρατίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, ήδη εξηγήσατε η ιστορία αυτή είναι αρκετά μακροχρόνια, της είχε και αρχικά ζητήσει αυτές Πολιτική κομισιών και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημοκρατισμού και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν το τι σημαίνει εδώ πέρα, θα διατρέξω έτσι κάπως γρήγορα τις ε, διαπραγματεύσεις και τους γύρους ε, και την ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Εξωτερικών. Η Κομισιόν ε, εισήγαγε μια καθαρά τεχνική τροπολογία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό για πέρσι, για τον ΦΠΑ, για να δοθεί αρκετή ευελιξία έτσι ώστε να μπορούν οι αρμόδιοι να κρίνουν που θα υπάρχει επιλεξιμότητα των φόρων ε, σε μέσα τα οποία χρηματοδοτούνται από την κοινότητα. Συμφωνούμε πλήρως εδώ πέρα με τις τροπολογίες και επιπλέον μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή το Νοέμβριο και μετά από την πρόταση της νομικής υπηρεσίας ε, του Κοινοβουλίου και το τι συνέβη με τα άλλα τρία χρηματοδοτικά μέσα αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε τροπολογίες έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί με την διαδικασία που λέγαμε παλιά της ε, Επιτροπολογίας να εξετάζει το μέσο αυτό και τα άλλα τρία μέσα, το μέσο για δημοκρατία και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από όταν όμως ε, τέθη η ενισχύ συνθήκη της Λισαβόνας δεν υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα οπότε έπρεπε να ε, προτείνουμε νέες τροπολογίες. Στις 3 Δεκεμβρίου συνεδρίασε η Επιτροπή μας, είχαμε ανταλλαγή απόψεων και ζητήσαμε από τους συναδέλφους να μας δώσουν μια εντολή διαπραγματευτική με το Συμβουλό και την Κομισιόν για να μπορέσουμε να έχουμε σύμφωνα με το άρθρο 290 πράξεις κάτ εξουσιοδότηση για την υιοθέτηση εγγράφων στρατηγικής σύμφωνα με το μέσο αυτό και άλλα μέσα. Η Επιτροπή μας έδωσε αυτή την εντολή και ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για τα τέσσερα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, δηλαδή το Χρηματοδοτικό Μουσείο της της Δημοκρατίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλα δύο δεν ε, ζητήσαμε λοιπόν να γίνει κάποια ψηφοφορία. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα. Μετά από δύο γύρους διαπραγματεύσεων υπομορφήν ε, τριμερούς διαλόγου υπό την ηγεσία του κύριου Μίτσελ από την Επιτροπή Ανάπτυξης κατέστη πως ούτε η Κομισιόν το Συμβούλιο είναι ανοιχτή σε μια δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου από το Κοινοβούλιο για τα έγγραφα στρατηγικής ε, στις πράξεις αυτές κατεξιοδότηση ούτε καν για το τμήμα εκείνο των ε, εγγράφων στρατηγικής που εμπίπτουν σε αυτά τα οποία το άρθρο 290 ορίζει ως πράξεις κατεξιοδότηση. Οπότε θα θέλαμε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση και ένας μηχανισμός ακριβώς για αυτό το κομμάτι εκείνο των εγγράφων και των ενδεικτικών προγραμμάτων που μπορούν να θεωρηθούν πράξη κατεξιοδότηση. Για να έχουμε μία ίση βάση και για τα τέσσερα μέσα και για να μπορεί να διαπραγματευτεί το Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει πως τώρα χρειαζόμαστε μια ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο γιατί έτσι και τα τέσσερα αυτά μέσα έχουν την ίδια τροπολογία. Και μετά θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Πιθανότατα μετά την ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα πάει στην Ολομέλεια του Ιουνίου για ψηφοφορία στην πρώτη ανάγνωση και μετά θα έχουμε έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων. Τώρα πλέον είναι με ένας αγώνας μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιών για το ποιος θα έχει το, ε, για το εάν θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να εξετάζει τμήμα αυτών των εγγράφων. Τι θα ψηφίσουμε λοιπόν σήμερα. Οι, τις αρχικές τροπολογίες που αφορούν την αρχική πρόταση της Κομισιόν με τις οποίες δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και μετά αποσύρουμε όλες τις τροπολογίες που εισήχθησαν πέρσι υπό το RPS, δηλαδή τις 4, 5 και 6 και αντικαθίστανται από τις 9, 10 και 11 για τις ε, πράξεις κάτω εξουσιοδότηση που είναι οι ίδιες ε, και για τα τέσσερα μέσα. Νομίζω αυτά, είχα, αυτά έχω για την ώρα. Ευχαριστώ, Μπραντνερ. Ε, η συγχύτρια έχει άδεια μητρότητας και αντικαθίσταται από τον κύριο Μπουτικόφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ την ε, Φραντσίσκα Μπράντερ και ευχαριστώ τον συνάδελφο που ε, συνέταξε αυτή την εισήγηση για τον χρηματοδοτικό μέσο δημοκρατίας και δικαιωμάτων. Επομένω δεν μένει τίποτα άλλο κατά τη γνώμη μου ότι θα πρέπει απλώ να συνεχιστεί αυτή η διαδρομή την οποία χάραξε η συνάδελφο. και με το κείμενο και με αυτές τις τροπολογίες για τις κατανάθεση πράξεις όσον αφορά αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα ε, συμπεριλαμβανομένου και του μέσου για την δημοκρατία και τη σταθερότητα ε, όσον αφορά τον τριμερή διάλογο όπως προαναφέρθηκε δεν ε, ευωδόθηκαν προσπάθειες να συμφωνήσουμε και ακούσαμε και αυτές τις ε, σκέψεις όσον αφορά τις ε, κατά παραγγελία χρήσης κάποιων μηχανισμών οπότε και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει η ψηφοφορία τον Ιούνιο για την πρόταση της δεν προχώρησε η κατάσταση με τον ε, τριμερή διάλογο και όπως ξέρετε εκκρεμεί το τι θα γίνει όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ελαφρών όπλων. Πάντως όπως προαναφέρθηκε ακόμη περιμένουμε η Επιτροπή και το Συμβούλιο να κατεβάσουν από κοινού μια δήλωση για το τι θα να κάνουν όσον αφορά αυτά τα ελαφρά όπλα. Ό,τι πρόκειται να χρηματοδοθεί με το μέσον IFS. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Α, ο κ. Γκάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις ε, συναδέλφους που υπέβαλαν τις δύο εκθέσεις να αναφερθώ σε δύο σημεία και θα θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις από την Κομισιόν στο ένα. Μιλάμε για το ΦΠΑ. Ε, τέθη τώρα το αίτημα τη παραπομπή σε, να διαγραφεί η παραπομπή σε φόρους, τέλη κτλ. Η ερώτηση μου να τι συνέπειες έχει αυτό η ΜΚΙΟ αλλά και τα πολιτικά ιδρύματα που είναι εκεί στις χώρες χρειάζονται την δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ και αλλιώς δεν θα μπορέσουν να χρηματοδοθούν πολλά από αυτά τα έργα. Οπότε το να λείπει εδώ πέρα η παραπομπή βοηθάει αυτό ή μήπως η Κομισιόν θα έπρεπε να δει τα της να πει δηλαδή ότι επί της αρχής δεν επιτρέπεται και δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ αλλά μετά να κάνει μια εξαίρεση γιατί τελικά οι ΜΚΟ και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται εκεί πέρα δεν θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα έργα γιατί δεν θα έχουν παραπάνω μέσα για να πληρώσουν από την τσέπη τους το, το ΦΠΑ. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το οποίο θέλω να αναφέρω, για μια έτσι συζήτηση μετά την πρώτη ανάγνωση στον τριμερή διάλογο της Επιτροπολογίας βλέπουμε πως αυτό το οποίο θέλει το Κοινοβούλιο για το πώς θα ασκήσει την επιρροή του στο μέλλον και πώς θα κάνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο φαίνεται πως θα ε, κανει το κοινοβουλευτικο ελεγχο πέσει σε τείχο, έχουμε χτυπήσει τείχο εναντί της, ε, της Κομισιόν και του, του Συμβουλίου. Θα πάνε δηλαδή όλα τα μέσα αυτά σε μία γραμμή μετά την πρώτη ανάγνωση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε μετά να συζητήσουμε εάν θα μπορούσαμε εμεί να σκίσουμε ε, κάποια επιρροή για το πώς θέλουμε να έχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λέζιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της ομάδας μου, της ΓΚΟΕ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις ε, προσπάθειες της για να έχουμε μια συμφωνία στον κοινοβουλευτικό έλεγχο των ε, εξωτερικών αυτών μέσων. Όπως ξέρετε η ομάδα μου η Γκουε ήταν πάντα κατά της συνθήκης Λισαβόνας μεταξύ άλλων και για το ότι ακριβώς χάναμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε τέτοιες περιπτώσεις. Οπωσδήποτε αλλού κέρδισε το κοινοβούλιο, αλλά κατά την άποψή μου νομίζω πως κερδίσαμε δυσανάλογα λίγα σε σχέση με την Κομισιόν και τις πράξεις αυτές ε, κατ' εξουσιοδότηση. Οπότε βλέπετε το τι γίνεται και με οτιδήποτε αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και οτιδήποτε αφορά το Συμβουλίο και την κυρία Άρστον. Οπότε υποβαθμιζόμαστε ως το μοναδικό δημοκρατικά έρετο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν δεν ενισχύεται αλλά αποδυναμώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε σχέση δε με τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα, με το μέσο για την παραγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουμε τις τροπολογίες της ηγετρίας και θα τις υπερψηφίσουμε για να υπάρχει πραγματικός δημοκρατικός έλεγχος. Όσον αφορά το ίδιο το μέσο εξακολουθούμε να το απορρίπτουμε λόγω του αντιδημοκρατικού του χαρακτήρα ο οποίος επίσης πλήττει την κυριαρχία χωρών και στην ε, τελική ψηφοφορία η δική μας η θέση θα είναι αυτή της εποχής Οπότε και στα υπόλοιπα μέσα θα υπερψηφίσουμε τις τροπολογίες αλλά στην τελική ψηφοφορία όπως σας είπα και πάλι θα ψηφίσουμε Ευχαριστώ. Στον κύριο Μενιέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη Διεύθυνση Ρελέξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με την τεχνική τροπολογία για τους φόρους. Πρόκειται για μια θα έλεγα τεχνικού τύπου ευθυγράμμιση με τα υπόλοιπα μέσα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους ήδη αυτό το στοιχείο θα έλεγα ευελιξίας σε σχέση δηλαδή με τη μη επιλεξιμότητα των διαφόρων τύπων φορολογίας. Τα χρήματα των φορολογουμένων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να πληρώνονται τελωνιακοί δεσμοί ή διάφορες άλλες μορφές φορολογίας. Αυτή είναι η βασική αρχή και δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε από το συγκεκριμένο κανόνα. Πρόκειται για ένα επιπλέον στοιχείο θα έλεγα ευελιξίας έτσι ώστε ο συγκεκριμένος εξουσιοδοτημένος διατάκτης να θεωρεί ότι είναι επιλέξιμο το τμήμα του ΦΠΑ για το τμήμα το οποίο αφορά συγκεκριμένες μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε χώρες ε, με τις οποίες δεν υπάρχει φορολογικού τύπου συμφωνία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαν παράδειγμα για μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρώσουν ΦΠΑ. Για κάποια περιφερειακά προβλήματα τα φορολογικά συστήματα είναι θα έλεγα ιδιαίτερος περιπλόκου αρχιτεκτονικής. Δεν δίδουμε λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση μια επιταγή εν λευκό, αλλά ρυθμίζουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Καλώς. Για να κλείσω. Ευχαριστώ συνάδελφε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα είπε ο κύριος Γκάλερ. Σωστά είπατε κύριε Γκάλερ πως το κοινοβούλιο πράγματι έχει χτυπήσει τείχο εναντί Συμβουλίου και Κομισιόν σε αυτά τα θέματα, αλλά και εμείς σκοπεύουμε να δείξουμε πως και εμείς είμαστε σκληροί εξίσου σκληρή αν θέλετε και θα αποφασίσουμε ανάλογα στον Ιούνιο στην Ολομέλεια πως ε, θα πρέπει και εμείς πλέον να συμπεριφερθούμε ανάλογα και όπως ε, μας αντιμετωπίζουν. Thank you. Uh, thank you, colleagues, for... Κύριε Γκάλ, ευχαριστώ. Θα απαντήσω μόνο στον κύριο Γκάλερ, αν κατάλαβα καλά. Συμφωνώ μαζί σας, πλήρως. Είναι πολύ σημαντικό για το έργο των ΜΚΟ εκεί πέρα να ψηφιστούν αυτές τις τροπολογίες και η Κομισιόν να αλλάξει την αρχική της πρόταση για να είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ. Και αυτό είναι σαφές και στην έκθεσή μας. Οπότε υποστηρίζουμε πλήρως αυτή την πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν. Αυτό το οποίο συνέβη εδώ και μπορεί ίσως να σας μπερδεύει είναι πως είχαμε δύο μέσα το DCI και το Μέσο για την Πρόοδο της Δημοκρατίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επειδή εμείς τα βλέπουμε αυτά σε δύο διαφορετικές ε, επιτροπές ε, είχαμε μόνο το ένα για εμάς και το άλλο βεβαίως της αναπτυξιακής ε, συνεργασίας ε, πήγε στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Αλλά η δική μας Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Κομισιόν για να τροποποιηθεί. Okay. Εντάξει, γιατί ήταν λίγο περίπλοκο. Ελπίζω να ήμουν σαφής. Okay, sorry. Uh, do I have to repeat? Να τα ξαναπώ. Α, λοιπόν. Υποστηρίζουμε την Επιτροπή με τον να συμπεριλαμβάνουμε την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ. Υποστηρίζουμε την Κομισιόν. Οπότε είναι σαφείς εδώ οι τροπολογίες. Μάλιστα, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Περνάμε τώρα στο σημείο 8, πρόταση ψηφίσματος ε, για την ε, αίτηση ένταξης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση αυτής της χώρας είναι σε πολύ ε, δύσκολη αυτή τη στιγμή μετά από την κατάρρευση του πιστοτικού συστήματος και τις προώρες εκλογές. Αυτή τη στιγμή στην εξουσία είναι ένας πολιτικός σχηματισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται φιλοευρωπαϊκός και η κυβέρνηση της χώρας αυτής αποφάσισε να καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας έτσι ώστε να διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Τον Φεβρουάριο του 2010 η Επιτροπή εξέδωσε θετική γνώμη. Το Συμβούλιο δεν έχει εξετάσει ακόμα τη συγκεκριμένη άποψη και το θέμα μπορεί να συζητηθεί στα πλαίσια της συνάντησης κορυφής του ενεστώτος μηνός. Ο κ. Πρέντα είναι ο εισηγητής, επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το Ρέικιαβικ και συναντήθηκε με ε, πολλούς ενδιαφέροντες παράγοντες της χώρας, την κυβέρνηση, του Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών υπέρ και κατά της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Πρέντα συζήτησε μαζί τους τα θέματα που άπτονται της υποψηφιότητας της Ισλανδίας. Ο εισηγητής ενέταξε στην έκθεσή του τις πληροφορίες τις οποίες συνέλεξε κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στην Ισλανδία και του ζητώ να πάρει το λόγο και να συμμεριστεί τις εντυπώσεις του μαζί μας. Και πέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως πολύ σωστά είπατε, την προηγούμενη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να συναντήσω στο Ρέικιαβικ τους ομολόγους μας της Ισλανδικής Βουλής. Συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Γεωργίας και Αλίας. Ενός τομέα πολύ σημαντικού για την Ισλανδία. Είχα επίσης την δυνατότητα να συναντηθώ με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που εκφράζονται υπέρ ή κατά της ένταξης της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επίσης και με τους συνδικαλιστές ηγέτες, τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών κτλ. Όλα αυτά ε, για να μπορέσω να κατανοήσω το σκεπτικό αν θέλετε της αίτησης ένταξης της Ισλανδίας που κατετέθη τον προηγούμενο Ιούλιο. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει μια θετική γνωμοδότηση και περιμένουμε στο άμεσο μέλλον και την άποψη του Συμβουλίου σχετικά με την πιθανή υποψηφιότητα της χώρας. Για την συγκεκριμένη έκθεση να σας πω ότι ξεκίνησα από κάποια συγκεκριμένα θέματα. Καταρχάς τα πολιτικά κριτήρια, όπως γνωρίζουμε όλοι, η Ισλανδία είναι μια χώρα με βαθύτατες δημοκρατικές παραδόσεις, υπάρχει ένας βαθύτατος υποδειγματικός θα έλεγα πολιτικός πολιτισμός στη χώρα. Τα περισσότερα συνεπώς από τα πολιτικά κριτήρια εκπληρούνται εκ των προτέρων. Όπως το υπογράμμισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Μας έχει ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά που αφορούν κυρίως ε, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τώρα για τα οικονομικά κριτήρια. Από τη μία Γνωρίζουμε ότι η Ισλανδία συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, κάτι το οποίο αποδεικνύει την ικανότητα της συγκεκριμένης χώρας να λειτουργεί ε, σε επίπεδο οικονομικό, επαναλαμβάνω, ανταγωνιστικά και να συμμετέχει στην ενιαία αγορά. Όπως γνωρίζουμε η χώρα αυτή κατατρίχεται τον τελευταίο τουλάχιστον καιρό από μια βαθύτατη οικονομική κρίση. Παρ' αυτά ε, υπάρχουν κάποια θετικά μηνύματα τα οποία υποδεικνύουν την δυνατότητα επιστροφής σε μια σταθερότητα οικονομική και από ό,τι φαίνεται η κατάσταση θα βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον. Στην Ισλανδία έχει ξεκινήσει μια πολύ έντονη συζήτηση για την έρευνα την οποία κάνει μια ad hoc επιτροπή για την οικονομική κρίση και την κατάρρευση ε, του πιστοτικού ε, ε, συστήματος της χώρας. Τα αποτελέσματα αυτής της Επιτροπής Έρευνας θεωρούνται στην Ισλανδία σαν βάση για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των εταίρων τους. Βλέπουμε ότι υπάρχει βέβαια μια γενικότερη έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην πολιτική τάξη της χώρας. Το ίδιο έγινε και στις τελευταίες εκλογές, όπου υπήρχε και ένα κόμμα εναντίον του συστήματος, το οποίο επευλήθηκε στις τοπικές εκλογές. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και άλλο ένα πρόβλημα, το οποίο είναι αρκετά ευαίσθητο είναι το θέμα των διμερών σχέσεων ανάμεσα στην Ισλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία, όπως επίσης και την Ολλανδία. Γιατί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μετά από την επιστολή την οποία έστειλαν στην κυβέρνηση της Ισλανδίας την προηγούμενη εβδομάδα και η κυβέρνηση είπε ότι θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τη Μεγάλη Βετανία και τις κάτω χώρες και ελπίζω εν πάση περιπτώσει το ταχύτερο δυνατό να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα της, Ευρω... της ε, Ισλανδίας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπα, η Ισλανδία ανήκει ήδη στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι η Γεωργία και η Ελία. Η Γεωργία και η Αλία σύντομα θα περάσουν από μια νέα διαδικασία μεταρρύθμισης βέβαια και γι' αυτό η Ισλανδία και τα υπόλοιπα φυσικά κράτη-μέλη στα πλαίσια ενός στενού διαλόγου θα καταλήξουν σε μια επικοδομητική λύση. Για τα θέματα της περιφερειακής συνεργασίας, στην έκθεσή μου επιμένω στον στρατηγικό ρόλο τον οποίο έχει η Ισλανδία. Όταν γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γιατί θα είναι το μοναδικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα ανήκει στη λεγόμενη περιαρτική ζώνη. Σε αυτή τη φάση το 33% των Ισλανδών είναι υπέρ της ένταξης της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η κατάσταση όπως είπα είναι ρευστή και όλα τα πολιτικά κόμματα με εξαίρεση τους σοσιαλδημοκράτες, ε, έχουν εσωτερικές διαιρέσεις γύρω από το θέμα της ένταξης. Επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ δημοκρατική χώρα, ανοιχτή στο διάλογο και ενθαρρύνω και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο αυτό και να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία έτσι ώστε όλες οι πλευρές ε, της Ισλαμικής κοινωνίας να μπορέσουν να εκφραστούν. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Η Προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 5η 3 Ιουνίου. Δεν έχουμε χρόνο. Και είναι απαραίτητο να υιοθετήσουμε το συγκεκριμένο ψήφισμα πριν από την συνάντηση κορυφής. Συνεπώς, προθεσμία κατάθεσης των απολογιών η 3η Ιουνίου στις 6 ε, το απόγευμα. Το λόγο έχει η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Ε, κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε στα περισσότερα με την κυρία Νταν Περέντα τον κύριο Αλλά ίσως είναι, τα παρουσιάζει κάπως θετικά τα πράγματα. Ναι, με ξέρει τι λέω και γελάει. Ε, λέει ο ίδιος πως όταν μιλάμε για την ένταξη της ε, Ισλανδίας δεν υπάρχει πολιτική συνένεση. Το λέει μόνος του. Πάντα έτσι ήταν. Και τώρα, έχοντας κατά νου την οικονομική κρίση, οι πολιτικές αρχές θέλουν να ενταχθούν στην Ένωση, αλλά ο λαός είναι διχασμένος. Οπότε αναρωτιέμαι, εάν πραγματικά είναι βάση αυτή ε, ένταξης μιας χώρας. Κατόπιν, κύριε Πρόεδρε, έχω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Παράγραφος 8. Η Ισλανδία έχει υποχρεώσεις στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί είναι τόσο θετικός ο Χριστιαν Ντανπρέντε. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ την προηγούμενη εβδομάδα η αρχή επιτήρησης απέστειλε επιστολή σύμφωνα με τη διαδικασία επί παραβάση για να τηρηθεί και να εφαρμοστεί η σχετική ε, νομοθεσία. Μιλάμε για το σύστημα εγγυήσεων καταθέσεων. Η 7, κύριε Πρόεδρε, κατά την αίσθησή μου, βλέπετε εδώ πέρα πως ζητάει εξηγήσει από την Ισλανδία. Οπότε πώς το αξιολογείτε. Και έχουμε εδώ πέρα την γνωμοδότηση της Κομισιόν, η οποία δεν είναι τόσο θετική όσο ο εισηγητής μας. Η δε συμβουλή της Κομισιόν είναι ότι όσον αφορά την αλληλεία, όσον αφορά τη γεωργία, όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, όσον αφορά το περιβάλλον, όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την επιτήρηση. Σε όλους αυτούς τους τομείς πρέπει να γίνει ακόμα σκληρή δουλειά. Πώς δεν έχουν ε, εκπληρωθεί αυτά τα οποία ζητάει ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Οπότε, Κριστιαν, νομίζω ότι παρά θετικός. Εγώ θα πήγαινα περισσότερο προς την επικριτική σκοπιά της Κομισιόν. Δεν έχω την αίσθηση πως την Σύνοδο Κορυφής ε, που έρχεται θα έχουμε συμφωνία για την Ισλανδία γιατί δεν έχουν και τη δυνατότητα να αποφασίσουν ε, κάτι τέτοιο αρκετέ κυβερνήσει. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. ECR συμφωνεί με την υποψηφιότητα που θα έπρεπε να έχει υποβληθεί και εγκριθεί νωρίτερα. Εάν επομένω ευοδοθεί αυτό το αίτημα, τότε αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο, καρότο ας πούμε, ούτως ώστε να μπορέσει και η Νορβηγία να ακολουθήσει την ίδια οδό. Η Ισλανδία γενικά είναι μια στέρεα σταθερή χώρα όμως τώρα περνά κάποια πάρα πολύ επικίνδυνη συγκυρία, μια που είχαμε αυτού του είδους την αμελέστατη διαχείριση των χρηματοοικονομικών που έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και της πτώχευσης. Και τώρα προσπαθούν να δουν πώς θα μπορέσουν να επαναδιαπραγματευτούν το χρέος του και να το αναδιαρθρώσουν κάτι το οποίο προχωρά παράλληλα με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως ξέρετε πάρα πολλοί Βρετανοί είχαν καταθέσει τραπέζι εκεί οπότε είχε εμπλακεί φυσικά πάρα πολύ ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και το ίδιο ισχύει και για τις ε, κάτω και όπως ξέρετε και στις ε, εκλογές τις Ολλανδικές πρόκειται επίσης να χρησιμοποιηθεί το σχετικό επιχείρημα κατ' δεν συνέβη στη δική μας χώρα. Πάντως, εμείς είμαστε φανδόν υπέρ της ένταξης της Ισλανδίας και επίσης όσον αφορά και την ρύθμιση του χρέους ε, το οποίο πρέπει φυσικά να ρυθμιστεί αλλά το βλέπουμε χωριστό θέμα σε σχέση με την ένταξη της χώρας. Και πάντως η βασική πρόκληση εδώ είναι το πώς θα πείσουμε τους Ισλανδούς για τα υπέρ της ε, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ε, να πιστούν και για τα θέματα αλίας που τους καίνε και ότι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους χορηγήσει κάποια παρέκκληση που γνώμη μου θα πρέπει να τους χορηγηθεί μια που βρίσκονται σε τέτοια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Δηλαδή, να μπορούμε να φέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νορβηγία και Ισλανδία χωρί η ένταξη να του σκοτώσει τον κλάδο τη ε, αλίας. είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί συζητούν ότι το έχουμε παρακάνει με τη διεύρυνση. Δεν νομίζω όμω ότι αυτού του είδου η, η, η επίκριση τη υπερβολή ούτω πριν τη διεύρυνση καλύπτει του ε, Σκανδιναβού αυτού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, ούτε θα υπάρξει πρόβλημα μετανάστευση, το οποίο να είναι αποκύημα αυτή τη διεύρυνση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριο Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όσο Ολλανδέζα που δεν έχω λογαριασμό στην iSave, συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει ο συγητή πως δεν πρέπει να εμποδίσουν οι διμερείς εξελίξεις το να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία. ε με, συγχωρείτε εδώ πέρα, με αφαιρέθηκα. Μου έστρεψαν αλλού την προσοχή. Να ξεκινήσουν λοιπόν οι διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία. για αυτά ε, δε τα οποία ρωτάει ο συνάδελφος για τις Ολλανδικές εκλογές. Όχι. Οι Ολλανδοί πολιτικοί προσπαθούν να κρατήσουν εκτός προεκλογικού αγώνα τα ευρωπαϊκά. Μιλάμε μόνο για την κρίση και μόνο για την κρίση στη χώρα μου. Ε, δυστυχώς. Αυτό το οποίο είναι κρίσιμο στην ένταξη της Ισλανδίας στην Ένωση και είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο ε, λέμε για τα Βαλκάνια όπου οικοδομείται η δημοκρατία. Η Ισλανδία έχει μία από τις αρχαιότερες δημοκρατίες και πρέπει να την επενέσουμε και βλέπουμε πως εκεί πέρα οι πολίτες παίρνουν τα δικαιώματά τους στα χέρια τους. Ειδικά να δούμε το τελευταίο δημοψήφισμα για την αποπληρωμή της Μεγάλης Βρετανίας και της Ολλανδίας όπου ψήφισε όχι ο πληθυσμός και βλέπουμε πως στήριξη του πληθυσμού για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ισχυρή. Δεν ξέρω νομίζω καλό είναι να γίνει δημοψήφισμα και για την ένταξη. Και αν θέλουν πράγματι να ενταχθούν, να τους προσκαλέσουμε. Και εάν πρέπει να ενταχθούν, πρέπει να δούμε και εμείς από την πλευρά μας τι θα κάνουμε. Έχει έναν αηφόρο τομέα αλίας από τον οποίο μπορούμε να διδαχτούμε και δεν μπορούμε να αφήσουμε εμείς τις τεράστιες στράτες μας να πάνε εκεί πέρα και να αδειάσουν τα νερά τους. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει επίσης με την ζώνη των 200 μιλίων ε, οικονομικής δραστηριότητας ε, που έχει η Ισλανδία και μιλάμε βέβαια εδώ πέρα για την αηφόρο όπως σας είπα αλληλεία. Επίσης σημαντικό είναι πράγματι να κάνει κάτι για την οικονομική επίβλεψη η Ισλανδία γιατί τα διμερεί ζητήματα πράγματι δεν πρέπει να εμποδίσουν την ένταξη, αλλά ίσως να φταίει ότι είμαι και Ολλανδέζα, θεωρώ επίσης πως πρέπει να κάνει κάτι να, να ξεκαθαρίσει εκεί πέρα τα του της, του δημοσιονομικού οίκου της η Ισλανδία και το χρηματοπιστωτικού. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Θα συμφωνήσω με την Ρία Όμεν Ρόιτεν αυτή τη φορά. Τα βλέπουμε πολύ θετικά τα πράγματα, κύριος Πρέντα, και το αποτέλεσμα των δημοσιονομικών, των χρηματοπιστωτικών συμφωνιών καταψηφίστηκε γιατί να συμβεί κάτι διαφορετικό τέτοιο τώρα. Μπορεί να θέλει ηγεσία αλλά ο λαός είναι κατά. Δεν είναι λοιπόν σωστό αυτό σε μια δημοκρατική Ευρώπη. Εγώ δεν θα ήμουν υπέρ πράγματι ενό δημοψηφίσματος εδώ πέρα. Κύριος Τάλερ. Στο ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω πως ε, υποστηρίζω την ένταξη της διαπραγματεύσης και την ένταξη της Ισλανδίας. Συγχαίρω εδώ πέρα τον κύριο Νταν για την πολύ καλή έκθεση. Βρήκαμε και στην Ισλανδία πράγματα τα οποία βεβαίως ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί τελείως και πρέπει να ξεκαθαριστούν πριν Έχουμε υπογραφές, οπότε σας ευχαριστώ για την ε, εκθέση αυτή. Ανησυχώ τώρα βεβαίως για τις παρατηρήσεις των δύο Ολλανδών συναδέλφων που σχετίζονται ίσως με τις εκλογές, αλλά ίσως να πηγαίνουν και παραπέρα από αυτό. Δηλαδή, τα διμερεί ζητήματα παίζουν ε, και θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εγώ θα πρότεινα στις επόμενες φάσεις, ε, θα αυτό προτείνω στον εισηγητή, σε αυτές τις περιπτώσεις να τίθεται μια προθεσμία στα κράτη για να λύνονται διμερώς τα προβλήματα π.χ. Ε, εντός 12 μηνών. Αλλιώς να πηγαίνουν στο Διεθνές Δικαστήριο. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση τι θα γίνει. Μικρά προβλήματα θα εμποδίζουν συγκεκριμένες χώρες να ενταχθούν. Και ένα Διεθνές Δικαστήριο μπορεί να αποτελέσει μία μέθοδος στην οποία θα μπορούσαμε να προσφύγουμε πριν κλιμακωθούν τα πράγματα θα ήθελα επίσης να ελπίζω πως ε, ναι, πράγματι το Συμβούλιο πρέπει να πει πως υπάρχει και μία ευθύνη εδώ πέρα και πρέπει να υπάρξει και ένας ρυθμός σε σχέση με την Ισλανδία γιατί έχει καταθέσει εδώ και καιρό αυτή την έτσι η Ισλανδία και σημαντικό είναι να δούμε τι θα γίνει με τις παγωμένες αυτές ε, διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις έπρεπε επίσης να ξεκινήσουν με την Ισλανδία και την ε, μου για να ολοκληρωθούν κάποτε. Κύριε Πρέντα, τώρα ήρθε η ώρα για σας να δευτερολογήσετε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους αδέλφους οι οποίοι έλαβαν τον λόγο, λέει ο κύριος Πρέντα όλους λοιπόν τους αδέλφους που είχαν την καλοσύνη να λάβουν το λόγο και να παρέμβουν τώρα όσον αφορά τα όσα ερωτήθηκαν ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικά πρώτα πρώτα κατά πόσον μπορεί είναι έτοιμη η Ισλανδία δεύτερον είναι, αυτό γίνεται στην σωστή χρονική συγκυρία είναι σοβαρά, πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα και η Ισλανδία δικαιούται να δώσει την απάντηση και ακριβώς αυτό θα ήθελα και να σας πω δεν θα απαντήσουμε εμείς αντί για την κυβέρνηση ή τους πολίτες της χώρας. Αυτοί θα μας πούν. Και αυτό θα γίνει δυνάμει του άρθρου 49 της συνθήκης που προβλέπει ότι κάθε χώρα στην Ευρώπη δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα. Τώρα, όσον αφορά το πνεύμα της ε, του, του, κειμένου μου. Βεβαίως και θα πρέπει κανείς να είναι θετικός με κάθε περίπτωση υποψηφιότητας για ένταξη. Και κατά τη γνώμη μου, τον Ιούνιο το Συμβούλιο θα αποφασίσει και θα πρέπει αυτό να γίνει αμελητή. Πάντως, ευχαριστώ τον κύριο Τάνοκ για τα όσα είπε, και επίση είναι πάρα πολύ εύστοχο το ότι συνέδεσε την προσφυγή τη Ισλανδία με την ενδεχόμενη προσφυγή τη Νορβηγία. Πρόκειται για θέματα τα οποία όλοι τα έχουν υπόψη τους. Επίσης ευχαριστώ για το όσα είπατε και για την αλία. Είναι θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει και άλλους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν σχετικά. Οι διαπραγματεύσει θα πρέπει να συνεχιστούν, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια λύση μακρόπνοη και να δούμε τι θα ακολουθηθεί στην πράξη σε σχέση με την Ισλανδική Αλληλιακή Αργεντινή και εσά σα ευχαριστώ. Μα μιλήσατε για δημοψήφισμα. Βεβαίω, προβλέπετε στη χώρα να γίνει δημοψήφισμα ε, όταν κάπου καταλήξουν οι διαπραγματεύσει. Τότε θα κληθεί ο λαός της χώρας να κρίνει και να αποφασίσει το τι θα γίνει. Ξέρετε, στη χώρα έχει κλείσει το θέμα. Θα γίνει δημοψήφισμα. Τώρα όσον αφορά με τη, την, την επίλυση της ε, χρηματοοικονομικής κρίσης που έχει χτυπήσει τη χώρα, βεβαίως και θα πρέπει αυτό κατά προτεραιότητα να αντιμετωπιστεί. Τώρα όσον αφορά την ΕΖΕΣ, επίσης Έχουμε ε, ε, τη σχετική τροπολογία. Όχι, όχι, όχι, δεν το ξέχασα. Απλώς θα πρέπει να γίνει συντονισμός του τι θα κάνουμε εδώ σε σχέση με την δημοσιοποίηση της ε, σχετικής επιστολής για το χρέος. Κύριε Σαντζεντίνη, έχετε δίκιο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την εμπειρία της χώρας. Επίσης νομίζω εκάλυψα τα υπόλοιπα τα οποία είπατε και σε σχέση και με, την, με το δημοψήφισμα αλλά και πάλι ευχαριστώ τον κύριο Τάνοκ για όσα είπε. Τώρα όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα για τις διμερείς επαφές δεν ξέρω αν ε, χρειάζεται ε, να τάξουμε τέτοια προθεσμία. Υπάρχει αυτό το θέμα για τι καταθέσει μεταξύ ε, κάτω χωρών, Ηνωμένου Βασιλείου και Ισλανδίας. Αυτό νομίζω το θέμα θα έχει κλείσει ε, πριν ε, τελειώσει η χρονιά. Νομίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα από όσα πολλοί πιστεύουν. Δεν νομίζω ότι αυτό θα βαρύνει δυσμενώς στην υπόθεση της ε, ένταξης της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, προχωρούμε στο σημείο παριθμών 5, ε, το οποίο αφορά τη συμφωνία πανεσδοχή μεταξύ Ευρωπαϊκής Συνότητας και Πακιστάν. Νίλσεν, ε, για τους πράσινους ε, είναι η έκθεση αυτή, την έχει αναλάβει η κυρία Νικόλ Κιλ Νίλσεν. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόκειται τώρα να γίνει για τρίτη φορά η σχετική συζήτηση. Το θέμα είναι της καθής μια που έγινε αυτή η ε, συνάντηση κορυφής. Και διαπιστώνω ότι έχουμε μία και μόνη τροπολογία η οποία έχει κατέβει εκ μέρους του κυρίου Πρέντα. Επ' αυτού θα πρέπει να σας πω ότι τα επιχειρήματα που έχουν προταχθεί δεν με έχουν πείσει. Λέγεται ότι η συμφωνία αυτή δεν θα κατοχυρώσει το δικαίωμα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω ότι επ' αυτού ε, ορθώς έχουμε επιφυλάξεις. Έχουμε κάποιους ε, ειδικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το έχουν ε, ασχοληθεί. Ε, δεν συμμετέχουμε στη Μεκτή Επιτροπή Ελέγχου Κοινοβούλιο και νομίζω ότι έχουμε διάφορα προβλήματα, διάφορες παραδιάσεις των δικαιωμάτων που έχουν διαπιστωθεί, ακόμα πάντως υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης και δεν έχω πιστεί για όσο λέτε κύριε Πρέντερ στην ε, τροπολογία σας. Συνεχίζω και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς όσον αφορά τον αγώνα μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην προηγούμενη Ολομέλεια ή στο Στρασβούργο από παντού άκουσα συναδέλφους που είπαν για τις επιφυλάξεις, για τη δυσαρέσκεια που νιώθουν όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Εις βάρος ε, μειονοτήτων θρησκευτικών, εις βάρος των γυναικών, ε, ήταν τα θέματα μας μας είχαν προσχωρήσει το ολομέλεια, οπότε και εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με όσα είπαν όλοι οι συνάδελφοι. για τη θανατική ποινή. Όταν έχει κυρώσει η χώρα τη νική της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Όλα αυτά ενδιαφέρουν τη συζήτησή μας και την εκθέσή μας και συνεχίζω να πιστεύω ότι ενώπιον μας έχουμε μία συμφωνία ελάχιστα ικανοποιητική. Άρα τα πράγματα μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν. Έχουμε 11 συμφωνίε που έχουν προηγηθεί, δεν έχει γίνει σωστή αξιολόγηση, αλλά θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση και θα πρέπει να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα πριν προχωρήσουμε στην έγκριση μιας νέας συμφωνίας, γιατί νομίζω ότι επιδέχεται σημαντικές βελτιώσεις αυτή η συμφωνία. Πάρα πολλά είναι φλού και αόριστα ακόμα. Τι γίνεται με την προθεσμία θέσεως ε, ισχύει. Τι γίνεται με τους ελέγχους της Μικτής Επιτροπής, τι γίνεται ε, με το ότι ε, δεν έχει ρυθμιστεί η αρμοδιότητα για την τακτοποίηση, τη ρύθμιση των προσφύγων από το Αφγανιστάν επομένω. Η κυρία Μάλουσον, η αρμόδια επίτροπο μπορεί να ασχοληθεί με αυτή τη συμφωνία και να τη βελτιώσει. Νομίζω ότι είναι εφικτό 100% και ε, το Κοινοβούλιο προς τιμή του καταψήφισε τη συμφωνία SWIFT. Γιατί θέλαμε περισσότερες εγγύσεις όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Άρα θα πρέπει να έχουμε συνεπή και αντίστοιχη στάση όσον αφορά τα δικαιώματα Αφγανών και Πακιστανών. Έχουμε επομένως ιστορική ευκαιρία για πρώτη φορά να τοποθετηθούμε στον αφορά τη Συμφωνία Πανεπιστοχής και μια ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε. Και καθ' αυτόν τον τρόπο να αποδείξουμε ότι μα ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να εξασφαλίσουμε τη βελτίωση της συμφωνία. Είναι θέμα αξιοπρέπειας και συνέπειας του Κοινοβουλίου. Και βεβαίω δεν μας ενδιαφέρει το ότι όλα αυτά είναι για το Πακιστάν. Για όποια χώρα και να εξαγγέλλονται κάποιες αρχές, ας πούμε ακόμα και η συνθήκη της Λισαβόνα. θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στο στον επεραμεινόμαστε των ιδιών μας και επόμενος αυτό θα πρέπει να γίνει που είπαμε με αυτήν τη συμφωνία που δεν είναι ικανοποιητική. Περιμένω τις παρατηρήσεις σας. Πρώτα πρώτα θέλω το λόγο κύριο Πρέντα. Στι προηγούμενε συζητήσει που κάναμε, Πρόεδρε, στην Επιτροπή μα, σα τα είπα. Σα είπα για ποιου λόγου θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει αυτήν την συμφωνία. Είχα κατεβάσει από εκείνο με τον κύριο Στράσε και μια τροπολογία. Και συνεπείς με τη γραμμή του ΕΛΚ είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο συνεργασίας επανεισδοχής με την χώρα αυτή. Επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Επίσης, θεωρώ ότι εάν τάξουμε κάποιες ε, προϋποθέσεις όπως παραδείγματος χάρη αυτούς τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής νομίζω ότι δεν είναι κάτι το βάσιμο μία τέτοια προϋπόθεση. Τώρα, όσον αφορά την συμφωνία. Μπορούμε τώρα να καλύψουμε τα όσα ορίζει το άρθρο 15 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ας μην έχει προσχωρήσει στη συνθήκη της Γενέβης. Θα πρέπει να τηρηθούν τα όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης και τα της μη επαναπρόθεσης. Και τα κρατημέλη πλέον αναλαμβάνουν την τήρηση αυτών των δεσμεύσεων. Δεν συμμετέχουμε στη Μεκτή Επιτροπή. Και αυτό γιατί οι ρυθμίσεις αυτές δεν είχαν γίνει πριν τεθεί σε ισχύ η συνδίκη της Λισαβόνας. Στο μέλλον μπορεί να καλυφθούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να διαφωνήσουμε με αυτή τη συμφωνία, να την, καταψηφίσουμε λόγω κάποιες ρύθμισης που είχε γίνει πριν στην συνθήκη της Λισαβόνας που τώρα βέβαια ισχύει πλήρω. Άρα, νομίζω ότι ο στόχο εδώ είναι κάτι το αναγκαίο. Αυτή η Συμφωνία Πανεγριστοχή είναι κάτι που μα έχει απασχολήσει πολύ καιρό και επομένω θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θα πετύχουμε περισσότερα εάν δεν πούμε όχι στη συνεργασία με αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος. Λόζινγκ. Ευχαριστώ. ήδη εξ ονόματος ε, της ΓΚΟΕ σε προηγούμενη συνεδρίαση σχολίασα τα συγκεκριμένα σημεία της ε, συμφωνίας. Σε ένα σημείο θα συμφωνήσω με την κυρία Κιλνίλσεν και εγώ ήθελα να πω πως πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να δούμε κατεπηγόντως τις πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τις θέσουμε να υπενθυμίσω επίσης πως ε, ειδικά η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις ασκούν κριτική σε αυτή τη ε, συμφωνία και μας προειδοποιούν να μην την υπογράψουμε. Τέλος, πρέπει να απορρίψουμε τις τροπολογίες πρέντα και ε, τη συμφωνία αυτή στο σύνολό της επίσης να απορρίψουμε. Αυτά και ευχαριστώ. Συγητής ε, για τα συμπεράσματα. Η συγητρία μας. Partenariat de coopération avec le Pakistan qui est en vigueur depuis 2004. Μιλάμε για κάτι το οποίο θα αρχίσει να ισχύει το 2014. 2004, συγγνώμη. Ε, κάτι το οποίο επομένως θα πρέπει να ε, το εξετάσουμε χωριστά σε σχέση με αυτό το οποίο σήμερα συζητούμε, ε, να δούμε ποιο είναι ο ρόλος τη χώρας όσον αφορά τη διεθνή καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας, διότι θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία που να λειτουργεί εύρυθμα. Βεβαίω και εγώ πιστεύω στην αποτελεσματική σχεδία Μάλμστρομ και γι' αυτό θα πρέπει τελικά να υπάρξει η ευκαιρία να κλειστεί αυτή η συμφωνία και ταυτόχρονα φροντίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία όπως μας είπατε ε, κατοχυρώνται από αυτή τη συμφωνία. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε ε, υπόψη τα όσα είπαν οι μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις. Και ας κάτσουμε να ρίξουμε μια ματιά στα όσα προβλέπει η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 7ης Μαΐου του 2010 και λέει ότι οι, εθνικοί φορείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν υποστηρίζουν από τις κυβερνήσεις, δεν ε, απολάβουν ανεξαρτησίας, ούτε έχουν ε, ισχύ, ούτε έχουν μάλλον αρμοδιότητα του να διεκπεραιώνουν ε, ατομικές καταγγελίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά είναι πρόβλημα. Οι δε αρχές που προστατεύουν τα δεδομένα ε, στην Ένωση δεν έχουν ερευνητική αρμοδιότητα, δεν έχουν ανεξαρτησία και σε 11 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει δυνατότητα του να, να, κάνουν τα περισσότερα αυτά που θα πρέπει να κάνουν. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανησυχία όσον αφορά το πώς θα γίνει ο έλεγχος ε, για την κατοχήρωση των δικαιωμάτων των ε, μεταναστών. Γι' αυτό και σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη συμφωνία επανεισδοχής και όλες τις άλλες που έχουν πράξει από διαπραγματεύσεις θα πρέπει να μνημονεύεται ποιος κάθε φορά είναι ο αρμόδιος από πλάση Ένωσης και Πακιστάν για να περιφρουρήσει τα δικαιώματα ε, των, προσώπων. Ευχαριστώ, λέει κύριε η ψηφοφορία θα ακολουθήσει στις 4.30 το απόγευμα. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι, δεν φαίνεται. Καλώς λοιπόν. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας. Μέχρι τις 11.30 διακόπτουμε. Α, για μια στιγμή, λάθο. Ο κύριο Μάιρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη μεγάλη σημασία που έχει η συμφωνία για μας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στην Ένωση. Υπάρχει ένας υψηλός αριθμός παράνομων μεταναστών που προέρχονται από το Πακιστάν. Μετά από μακρόχρονες διαπραγματεύσεις, ξεκινήσαμε θυμίζω στα τέλη του 2000 όταν πήραμε την εντολή μας. Πετύχαμε στο τέλος των διαπραγματεύσεων αυτό να καταλήξουμε σε μια εξισορροπημένη θα έλεγα απόφαση. Η συμφωνία αυτή έχει πολύ μεγάλη περιφερειακή σημασία στα πλαίσια της καταπολέμησης της ε, παράνομης μετανάστευσης. Εδώ έρχονται και οι διαπραγματεύσεις που γίνονται με την Τουρκία. Στόχος της συμφωνίας αυτής είναι η βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στις διοικήσεις των χωρών εκκίνησης και των χωρών υποδοχής. Είναι ένα αυστηρά διοικητικό μέσο, δεν αντιμετωπίζει το θέμα του καθεστώτος των συγκεκριμένων ε, προσώπων, ατόμων, τα θέματα των δικαιωμάτων του σαν παράδειγμα αντιμετωπίζονται από άλλα νομοθετικά μέτρα και μέσα. Αναγνωρίζουμε ότι το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο. Αξιολογούμε ότι και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και εσείς ζητάτε να ληφθεί υπόψη. Να υπενθυμίσουμε όμως πάντα ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες επηρεάζονται από τους παράνομους μετανάστες από το Πακιστάν με την βοήθεια ανθρώπων που ασχολούνται με το τράφικινγκ. Και νομίζω ότι η συμφωνία αυτή ε, στέλνει ένα μήνυμα προς αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με ε, το εμπόριο αυτό. Εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε και για τις άλλες συζητήσεις τις οποίες έχουμε και διαπραγματεύσει σύμφωνα με τη συνθήκη. Ε, σας ευχαριστώ που θα προωθήσετε, είμαι βέβαιο τη συγκεκριμένη συμφωνία η οποία μας πήρε πάρα πολύ χρόνο να την επεξεργαστούμε. Καλώς επαναλαμβάνω, σε 10 λεπτά θα